κάποιο ασυμβίβαστο με τα καθήκοντα του Ευρωβουλευτή. Ο κύριος Godfrey Bloom φεύγει από την ομάδα EFD με ισχύ από 9 Ιανουαρίου 2014 και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους. Το ΕΛΚ, οι Σοσιαλδημοκράτες και